Τώρα μένει μια έκθεση της κυρίας Ούρσουλας Γκάτσεκ για τα προβλήματα και προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Το λόγο έχει συγκίτρια για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, με μεγάλη χαρά παρουσιάζω την έκθεση αυτή για τα προβλήματα και τις προοπτικές Τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια που εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή ΕΛΕΦ τον περασμένο μήνα. Η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια δεν αντικαθιστά, που υποκαθιστά την εθνική. Είναι μια πρόσθετη αξία για τον Ευρωπαίο πολίτη και του δίνει πρόσθετα δικαιώματα όχι μόνο κυκλοφορία, αλλά και προξενικής προστασίας αναφορά στο Κοινοβούλιο και στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Η έκθεση του Κοινοβουλίου λαμβάνει υπόψη της την ε, έκθεση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια από, που κάλυπε την περίοδο από την 1η Μαΐου 2004 μέχρι 30 Ιουνίου 2007. Ήταν μια ξεχωριστή περίοδος αυτή γιατί πριν από 5 χρόνια 10 χώρες μέλη νέα έμπαιναν στην Ένωση. Η έβρινση μέχρι τότε δεν είχε ξαναγίνει τέτοιου, τέτοιας κλίμακας. Οι πολίτες των νέων αυτών χωρών άσκησαν τα δικαιώματά τους αμέσως, ιδιαίτερα της ελεύθερης κυκλοφορίας, του δικαιώματος να μορφώνονται εκτός, έξω από τη χώρα τους και άλλα. Αλλά η κλίμακα των μεταναστεύσεων έθεσε προβλήματα σε πολλές χώρες και για τις κεντρικές και για τις τοπικές αρχές. Οι τοπικές αρχές ιδιαίτερα όποτε είναι υπεύθυνε για υπηρεσίες στέγασης, υγειονομικές υπηρεσίες και παιδείας αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα με, τη νέα, με το νέο ρεύμα νέων μεταναστών. Έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μπορέσουν να υποφεληθούν και οι καινούργοι κάτοικοι των παλαιών χωρών από τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν και οι παλαιοί. Αλλά παρέμεινε κάποια άνηση μεταχείριση, καμιά φορά γιατί ο νόμος είχε ελλείψεις άλλες φορές γιατί δεν εφαρμοζόταν πλήρως. Η Επιτροπή ΕΛΕΦ ε, πήγε μια προσέγγιση, έκανε μια προσέγγιση πιο ρεαλιστική θέλησε να ταυτίσει τα προβλήματα δικαιωμάτων ενεργά θα διασφαλίζεται ιδιαίτερα και σε σχέση με την έγκριση της, Ευρωπα... της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας για την ελευθερία κυκλοφορίας των Ευρωπαίων πολιτών από τα κράτη-μέλη. Οι ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν για ε, την... Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανήκουν στις προτεραιότητες αυτού του έργου επικοινωνίας και ενημέρωσης. Υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εκστρατεία αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μέτρα καινοτομία ε, για την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των πολιτών να μεριμνήσουν, να, να ληφθεί μέρημνα ώστε θα συμμετάσχουν οι πολίτες σε αυτές τις ευρωεκλογές και να ζητηθεί από τους πολίτες να κάνουν πραγματική χρήση του δικαιώματος του εκλέγην και να συμμετάσχουν στις εκλογές. Συμβαίνει τούτο και θέλω ιδιαίτερα να το επισημάνω ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθημερινά να αποκτά σάρκα και οστά και να είναι αντικείμενο το οποίο θα χρησιμοποιούν οι πολίτες. Και τούτη η Ευρωβουλή και όλα τα 27 κράτη-μέλη και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα εθνικά κοινοβούλια και οι δημοτικές αρχές, δήμοι και κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι και όλες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση και άσκηση των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Χαίρομαι λοιπόν για το γεγονός ότι έγκαιρα πριν από τις Ευρωεκλογέ 2009 αυτή η έκθεση που δημοσιεύεται, δημοσιοποιείται από την κυρία Γκάτσεκ εμπλέκει αρκετούς από αυτούς τους σημαντικούς εταίρους που όλοι θα έπρεπε να οδηγήσουν στην ευδοκίμηση αυτής της ε, έννοιας της ηθαγένειας του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος των πολιτών. Είναι κοινό έργο όλων και πρέπει όλοι ως καθήκον να το δούμε ώστε η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι κάτι συμβολικό μόνο αλλά να το εννοούν οι πολίτες ως ένα χειροπιαστό συγκεκριμένο δικαίωμα στην καθημερινή ζωή το οποίο μπορούν να ασκήσουν ασκήσουν και να χρησιμοποιήσουν και πρέπει να το κάνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση έληξε. Αύριο 2 Απριλίου θα ξεκινήσουμε στις 9 η ώρα το πρωί και έχουμε δύο συνεδριάσεις. Ελίεται οι συνεδρίες. Καλό βράδυ.